Λοιπόν, νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προσέλθει ακόμα όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Φαντάζομαι ότι πρέπει πολλοί κόσμος ακόμη να, ξεχωρα... να ξεκουραστεί από την κουραστική ψηφοφορία που είχαμε σήμερα το πρωί. Θα έρχονται όμως, καθώς θα συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Ε, το ίδιο ισχύει βεβαίω και για την ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Τι έχουμε σήμερα. Κοινή ανταλλαγή απόψεων και συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για το Euronews. Να, να καλωσορίσω βεβαίως του συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού εδώ και χωρίς περαιτέρω ε, χρονοτριβή θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία ε, Γκρέσλε, την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού για να κάνει κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει και τους προσκεκλημένους μας και στη συνέχεια εγώ θα αναλάβω το συντονισμό της συζήτησης. Σας ε, καλωσορίζω κυρία Γκρέσλε και χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε σήμερα και οι δύο εδώ και μπορούμε να συμπροεδρεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευελιξία που έχει επιδείξει η Επιτροπή Πολιτισμού Εμάς μας απασχολεί η καταγγελία των εργαζομένων ε, του Euronews ε, σχετικά με ε, παρεμβάσεις του νέου ιδιοκτήτη του Euronews. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το Euronews με χρήματα ύψους 25 εκατομμυρίων το ευρώ το χρόνο αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις, γι' αυτό χαίρομαι που είναι μαζί μας και ο κύριος Πέτερς, ο διευθυντής του Euronews και ο κύριος Γκαριμπέρτη που είναι πρόεδρος της συντακτικής ε, επιτροπής του Euronews και ε, χαίρομαι που είναι μαζί μας και ο κύριος Αμπαμόντε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τοποθετηθεί και εκείνος. Έχουμε πραγματικά να κάνουμε με βαρύνουσες καταγγελίες διότι ε, οι συντακτικές και δημοσιογραφικές παρεμβάσεις ε, των ε, ε, συμμετεχόντων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να τύχουν τις προσοχής μας και γι' αυτό πρέπει και να γίνει σήμερα αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Πέτερς προκειμένου να μας παρουσιάσει τα πράγματα από τη σκοπιά του Euronews. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ για να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για την κατάσταση στη Euronews. Όπως κατάλαβα μετά την εισαγωγή της κυρίας Πρόεδρου, ήδη μας κατηγορείται για παρεμβατικότητα, κάτι που θεωρώ απαράδεκτο. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στην Euronews και θα σας εξηγήσουμε με μεγάλη μας ευχαρίστηση πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα και πώς λειτουργεί η Euronews αυτή τη στιγμή. Πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες για την Euronews. Πολλά από αυτά ήταν σωστά, άλλα ήταν λάθος. Περιέργως ε, λένε πολύ δεν γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση στην Euronews και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας διαφωτίσω λίγο για το που βρισκόμαστε και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στην εταιρεία μας. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από την αρχή. Το όραμα της επιχείρησής μας, ε, τι υποστηρίζουμε, τι προσπαθούμε να επιτύχουμε καθημερινά μαζί με όλους μας τους μετόχους, μαζί με, την, ε, πλειοψηφούσα, με το πλειοψηφούνα μέτοχο, τη Euroservice προσπαθούμε να παρέχουμε μια καθολική εμπειρία ειδήσεων, γνώσεων και πολιτισμών μέσω τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό μα DNA, γνωρίζοντα ότι η πολυμορφία προέρχεται από την αρχή ενωμένη στη διαφορετικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωση. και πιστεύουμε όλοι ακράδαντα και εγώ προσωπικά ότι ο ρόλος των μέσων μαζική ενημέρωσης δεν είναι να επηρεάζει τις απόψεις των ανθρώπων, αντιθέτως να τους ενδυναμώνει, να τους χειραφετεί. Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωση, είναι να χειραφετεί του ανθρώπους, να τους δίνει τα κλειδιά που τους βοηθούν να σχηματίσουν τη δική τους άποψη. Αυτό θέλουμε να, γίνεται, να κάνουμε εμείς και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μέσω ανεξάρτητων, ε, δεσμευμένων και αξιόπιστων ειδήσεων. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά στη Euronews. Το τελευταίο μας όραμα, ο τελευταίο μας στόχος είναι να κάνουμε τη Euronews έναν οργανισμό που θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επιρροή ε, από τη σήμερα σε ευρωπαϊκά θέματα. Και θα σας εξηγήσω πώς ακριβώς ε, επιθυμούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Λοιπόν, μερικά στοιχεία καταρχάς. Ε, θα γνωρίζετε ήδη πολλά για το Euronews, αλλά θα προσπαθήσω να σας συνοψίσω σε τέσσερις διαφάνειες τα βασικά στοιχεία. Το πρώτο, σήμερα εκπέμπουμε σε πάνω από 400 εκατομμύρια ε, σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβάνονται 300 εκατομμύρια ε, σε πλήρες ε, σε full time βλέπετε την κατανομή των διαφορών τμήματων της Euronews εδώ και βλέπετε ότι η Euronews είναι το πρώτος διεθνής σταθμός που μεταδίδεται στην περιοχή EMEA. 288 εκατομμύρια άνθρωποι είναι συνολικά η, ε, το κοινό της Euronews κάθε μήνα. 147 εκατομμύρια βλέπουν τη Euronews live και σε VOD σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ε, σε τηλεόραση και ψηφιακά την εβδομάδα και 40 εκατομμύρια την ημέρα. Θα δείτε εδώ, μπορείτε να δείτε εδώ την ε, κατανομή μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον. Έχουμε τους θέατες της τηλεόρασης. Ε, το ψηφιακό κοινό δεν είναι ακόμα αρκετά ισχυρό κατά την άποψή μας. Πρέπει να το αναπτύξουμε ε, στο μέλλον. Η Γερόνιος ε, απασχολεί περίπου χίλιους υπαλλήλους, από αυτούς 600 δημοσιογράφους, από περισσότερες από 30 υπηκότητες σε 13 γλωσσικές εκδόσεις. Έχουμε 8 γραφεία σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους ε, ε, ιδιοσιογραφικού πρακτορείου στις Βρυξέλλες. Να σας μιλήσω τώρα λίγο για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς στη Euronews αλλά ουσιαστικά και σε όλους ε, τους σταθμούς ε, μέσω μαζικής ενημέρωσης στον τομέα. Πρώτον, έχουμε ένα υπερβολικά ανταγωνιστικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο ε, εμφανίζεται, ε, εμφανίζονται ένα έω πέντε σταθμοί νέοι. Είμαστε πάνω από 250 δημοσιογραφικοί σταθμοί αυτή τη στιγμή. Οπότε η πίτα ε, της διαφήμισης ε, παραμένει ίδια και μάλιστα παρουσιάζει κάποια μείωση, οπότε το μερίδιο της πίτας για τον καθένα μειώνεται. Επίσης υπάρχει μεγάλη αλλαγή στο εικόνα που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το ψηφιακό κόσμο τώρα και με τους καταναλωτές να αναζητούν να ειδήσει με διαφορετικά άλλο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο και αυτά τα δύο κριτήρια έχουν ως αποτέλεσμα έναν κόσμο με υπερβολικά πολλές πληροφορίες ε, όπου ε, πρέπει ο καθένας να κάνει κάποια επιλογή. Ε, βλέπουμε την ίδια επανάσταση που χαρακτήριζε τη μουσική βιομηχανία πριν από 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα επιχειρηματικά μας μοντέλα, διότι κανένας από του συναδέλφου μα δεν έχει κάποιο μοντέλο που να λειτουργεί άψογα. Αν δείτε τον ανταγωνισμό, βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε χρόνο τίθεται το ζήτημα των ε, μέσων που χρηματοδοτούνται με μετοχές και επίσης βλέπουμε ε, ε, το, την Guardian, το New York Times, την Al Jazeera μέσα που αφορούν όλους τους τομείς ε, και βλέπουμε περικοπές ε, του κόστους ε, σε όλα αυτά τα μέσα και ποια είναι τα αποτελέσματα λοιπόν. Ο πρώτος στόχος είναι να παρέχουμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή προοπτική. Θεωρούμε ότι στο DNA της επιχείρησης έχει εγγραφεί ότι κάθε μέτοχος έχει δεσμευτεί για αυτό το στόχο, κάθε μέλος του προσωπικού της Euronews έχει δεσμευτεί για αυτό το στόχο και πιστεύουμε ότι η Euronews θα ευδοκιμήσει σε αυτό το ε, κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης λόγω του ισχυρού της και μοναδικού της DNA. Φυσικά ε, πιστεύουμε ακραδάντα ότι αν ε, χάσουμε την πολυγλωσία που είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό θα χάσουμε ε, ένα μεγάλο μέρος του κοινού μας με καταστρεπτικές επιπτώσεις για τα εισοδήματά μας και για τη θέση μας στην αγορά. Ε, αυτονομία, φυσικά ανεξαρτησία, αυτό αποτελεί ε, το βασικό θεμέλιο των δραστηριοτήτων μας και έχουμε τη διακυβέρνηση της επιχείρησης που προσπαθεί να τηρεί την ανεξαρτησία του μέσου αυτού. Όπως είπα, η πολυμορφία επίσης είναι ένας από τους ισχυρότατους στόχους μας Ίσως γνωρίζετε ότι ε, το βασικό μας αξίωμα είναι να εκφράζουμε, να παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις, την πολυμορφικότητα, την πολυμορφία των απόψεων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Για να δείξουμε ακριβώς την ευρωπαϊκή ταυτότητα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται η αντιπαραβολή των διαφόρων απόψεων ε, ε, ώστε να σχηματίζει το ευρωπαϊκό κοινό τη δική του άποψη ο τελευταίος στόχος, η τελευταία πρόκληση είναι η βιωσιμότητα. Όπως ε, είπα υπάρχουν πολλά σταθμοί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλές δυσκολίες οικονομικές, έχουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί ικανοποιητικά αυτή τη στιγμή, πρέπει να το επανασχεδιάσουμε πλήρως. Ο επανασχεδιασμός αυτός του επιχειρηματικού μας μοντέλου απαιτεί ε, αναδιοργάνωση, ανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής των ειδήσεων και αυτό αποτελεί στόχο ενός μεγάλου στρατηγικού σχεδίου που έχουν ψηφίσει οι, οι μέτοχοι πριν από την έλευση του Euronews Next ε, που θα κάνει μια επανάσταση ουσιαστικά στην Euronews. Θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Ε, κάτι άλλο που βοηθά στη βιωσιμότητα ε, σήμερα στην αγορά είναι η κλίμακα βρισκόμαστε σε ε, μια εποχή συγκέντρωσης ε, ε, το CNN αγοράστηκε από την Time Warner, η Sky από την Fox και εμείς είμαστε ένας μικρός οργανισμός που αντιμετωπίζει πρόβλημα ανταγωνισμού με γίγαντες και ένα από τα κλειδιά που πιστεύω εγώ θα μας βοηθήσει να ευδεικνύσουμε σε αυτό το περιβάλλον θα είναι να γίνουμε μεγαλύτεροι διότι χρειάζεται κανείς αυτή την κλιμακουσία ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Ας μιλήσουμε τώρα για τους μετόχους. Είναι ε, ένα από τα βασικά σημεία στα οποία ήθελα να εστιαστώ. Ε, η Media Globe Networks ε, κατέχει το 53% των, του μετοχικού κεφαλαίου της Euronews και οι δημόσιοι μέτοχοι κατέχουν το 47%. Όπως θα ξέρετε, εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε με ένα νέο ε, πιθανό εταίρο ε, μεταξύ των μετόχων της Euronews την NBC Universal ε, τον οργανισμό αυτό μέσω μαζικής ενημέρωσης που, με την οποία διαπραγματευόμαστε εδώ και ένα χρόνο περίπου Υποθέτω ότι και εδώ θα έχετε να κάνετε πολλέ ερωτήσει και επειδή δεν έχω χρόνο θα προσπαθήσω να σα παρουσιάσω συνοπτικά τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με αυτό. Ο στόχο είναι απλό. Η NBC θέλει να επεκταθεί διεθνώ έχει κατανοήσει ότι η Ευρώπη είναι μια βασικότατη αγορά για διεθνή επέκταση. Η NBC εκτιμά το γεγονό ότι η θέση των Αμερικανικών μέσων ουσιαστικά έχει καταληφθεί πλήρως από το CNN στην Ευρώπη και δεν θα μπορούσαν ποτέ να νικήσουν το CNN σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό το λόγο ήρθαν σε εμά προσπαθώντας να επιτύχουν κάποια ε, εταιρική σχέση στην οποία θα φέρουν αυτοί, θα συμμετέχουν με τον επαγγελματισμό τους, με την εμπειρία τους ε, που θα συνδυαστεί με τη δική μας εμπειρία και την τεχνογνωσία της Euronews στα ευρωπαϊκά θέματα. Ε, συζήτησα μια στρατική ξεκινώντας πριν από 1,5 χρόνο, ε, που θα απαιτήσει πολλή εμπειρία στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε εμεί και πιστεύουμε ότι η NBC θα είναι σημαντικό εταίρο που θα μα βοηθήσει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επιρροή από τη σήμερα. Και φυσικά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, αυτό το θέμα και να μου κάνετε και ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή συζητάμε με την NBC να αγοράσει το 25% των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Euronews και η Media Club Networks θα είναι στο 60% και οι δημόσιοι ε, μέτοχοι στο 15%. Αυτή η μείωση των δημοσίων μετόχων έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω φαντάζεστε. Και είναι σαφέ ότι οι Ευρωπαίοι δημόσιοι μέτοχοι δεν θέλουν ή δεν έχουν τα μέσα να υποστηρίξουν την Euronews οικονομικά πλέον. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό για μας και για αυτούς εφόσον συμφωνηθεί αυτή αφόσον καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία να μειωθεί το ποσοστό αλλά να διατηρήσουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι δημοσιομετοχοί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι η Euronews έχει δύο ε, εξουσίες ελέγχου ε, την πλειοψηφία των μετοχών που και τους δημόσιους μετόχους που έχουν έλεγχο ε, των, ειδήσεων και ο σκοπός είναι αυτός ο έλεγχος των ειδήσεων να παραμείνει στα χέρια των δημοσίων μετόχων οι οποίοι θα είναι και θεματοφύλακες του ναού όπως λέμε μερικές φορές για την ανεξαρτησία των ειδήσεων στην Euronews και για την ευρωπαϊκή αυτή αποστολή υπερασπίση των γενικών συμφερόντων της Ένωσης. Τι διασφαλίσει έχουμε ε, θέσει για να το σκοπό αυτό για να διατηρήσουμε την αποστολή γενικού ε, ενδιαφέροντος της Euronews ε, ε, είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης ανεξαρτησία στις ειδήσει της Euronews η ανεξαρτησία της σύνταξη είναι το πιο σημαντικό μας πλεονέκτημα, το πιο πολύτιμο μας πλεονέκτημα. Οπότε είτε ε, η NBC είτε ο πλειοψηφόν μετόχος είτε και εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία ε, των καταναλωτών της Euronews ε, βλέπουν Euronews λόγω της ανεξαρτησίας της και της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Αν χάσουμε αυτό θα χάσουμε την Euronews και θα χάσουμε την αξία της εταιρεία. Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι η αξία της εταιρείας ε, έγκυται σε αυτή την αποστολή της ε, γενικού ε, συμφέροντος και ανεξαρτησίας. Ο δεύτερος λόγος για αυτή την αποστολή είναι και ο θεμέλιος λήθος της σχέσης μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους δημόσιους μετόχους αλλά και για την MBC και, την... και τον μεγαλύτερο μας μέτοχο την Media Club Networks. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο με δύο ε, εποπτικά συμβούλια. Ένα εποπτικό συμβούλιο, το Supervisory Board, που επιβλέπει την ε, διαχείριση της επιχείρησης. Αυτό το εποπτικό συμβούλιο ελέγχεται από την Agips OS. Ε, και μετά έχουμε και το συντακτικό συμβούλιο που ελέγχεται από τους δημόσιους μετόχους και ο πρόεδρος αυτού του Συμβουλίου ε, έχει από κάτω 10 μέλη, 7 από τα οποία ε, ορίζονται, ε, διορίζονται από τους δημόσιους μετόχους και 3 από την ΑΚΙΜ. Αυτό το συντακτικό συμβούλιο ελέγχει το συντακτικό κομμάτι της Euronews, την αποστολή της που αφορά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και εποπτεύει την συντακτική ε, Διευθυντική Επιτροπή η οποία εποπτεύει τον ε, ε, Διευθυντή Ειδήσεων. Το τελευταίο κομμάτι που θέλω να αναφέρω είναι οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ειδικότερα με την DigiConnect, η οποία εστίασε ιδιαίτερα την προσοχή της στην πιθανή αυτή συμφωνία με την MBC καταλήξαμε σε κάποιες γραπτές δεσμεύσεις που αποτελούν κομμάτι του ε, εισπολιτού συμφωνίας ε, πλαίσιο που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη δέσμευση είναι να δεσμευτούμε ε, για αμεροληψία και στην ενημέρωση και ανεξαρτησία στην ενημέρωση επίσης. είναι μια αμοιβαία δέσμευση της Euronews ε, και της NBC Universal να υπερασπίσουμε αυτές τις βασικές υποκείμενες αρχές. Σκοπός είναι ότι τις πρώτες εβδομάδες μετά την άφηξη της NBC θα ε, καθορίσουμε ένα όραμα, ένα κοινό όραμα που θα είναι δημόσια έγγραφα μερικών σελίδων που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Euronews και που θα δημοσιευτούν παντού όπου η Euronews και η NBC αμοιβαία θα αναλάβουν δεσμεύσεις προς την Ευρω... όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αποστολή ε, Γενικών ε, Συμφερόντων της Euronews. Ε, δεύτερον, οι συντακτικές αρχές, οι συντακτικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης και η εξωτερική αξιολόγηση των ανεξάρτητων οργανισμών θα συνεχίσουν να ισχύουν. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει έλεγχος από τους δημόσιους μετόχους και θα εξακολουθεί να υπάρχει ο ίδιος έλεγχος Τη σύνταξη ε, στην Euronews. Η τρίτη δέσμευση είναι ότι θα διατηρηθεί η πολυγλωσία στην Euronews ε, διότι αποτελεί ένα από τα σημαντικά της πλέον εκτήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σα εξηγήσω ένα πράγμα που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Η Euronews ε, μεταδίδεται σε 13 γλώσσες σήμερα. Από αυτές έχουμε έξι βασικές γλώσσε, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά και ρώσικα τι σημαίνει αυτό, ότι αυτές οι γλώσσες ε, χρηματοδοτούνται αυτόματα, ε, χρηματοδοτούνται από την ίδια την Euronews και από κάποιον εξωτερικό εταίρο. Και μετά έχουμε τις άλλες γλώσσες, ε, ουγγρικά, ελληνικά, πορτογαλικά, αραβικά, φαρσί, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τουρκικά, που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Τηλεόραση της Τουρκίας και ουκρανικά, για τα οποία έχει πάψει πλέον η χρηματοδότηση. Όλες αυτές οι ε, ε, γλώσσες ε, χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένου εταίρους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συμβάσεις με πελάτες, με εταίρους. Και εάν ο εταίρο αυτό αποφασίσει να καταγγείλει τη σύμβαση, η Euronews αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μόνη της τις γλώσσες αυτές. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια σημαντική διευκρίνηση που θα έπρεπε να γνωρίζετε. Η τέταρτη δέσμευση είναι ότι η συμφωνία με την NBC Universal δεν θα οδηγήσει σε μειώσει του προσωπικού λόγω αλλαγέ στο μοντέλο παραγωγή. Ήδη μελετάμε ένα σχέδιο ε, ανασχεδιασμού. Ε, πρέπει να ξα... ανασχεδιάσουμε, όπω σα είπα, τον τρόπο παραγωγή ειδήσεων. Βρισκόμαστε εν μέσω αυτού του σχεδίου. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε με την NBC και η NBC δεν έρχεται εδώ για να κάνει περαιτέρω περικοπές ε, δαπανών. Αντιθέτως με τα χρήματα με το οποίο θα συμβάλλει η NBC στο, κεφάλαιο, στο μετοχικό κεφάλαιο της Euronews θα έχουμε περισσότερους πόρους ειδικότερα στον τομέα της συλλογής ειδήσεων με ε, την ιδέα για παράδειγμα να έχουμε μόνιμους απεσταλμένους σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες ε, της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. Η πέμπτη δέσμευση είναι ο βασικός ε, υπεύθυνο για το περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τα θέματα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λιούκ είναι μαζί μας εδώ ε, εκείνο είναι ο αρμόδιος για το περιεχόμενο του Euronews και σε όλες τις διαφορετικές συμφωνίες ε, υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις ότι αυτός ο υπάλληλο θα πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις του, την αποτελεσματικότητά του, τις δεξιότητές του για το ρόλο αυτό που θα παίξει και δεν θα είναι αντιευρωπαϊστής, θα πρέπει να είναι ένας πολίτης φυσικά μιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία δέσμευση είναι ότι το όνομα Euronews θα παραμείνει και θα εμφανίζεται. Ε, το όνομα μπορεί να γίνει βέβαια Euronews NBC, θα συνδυαστεί με το NBC, αλλά το Euronews θα είναι πρώτο και θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση ε, στην νέα επωνυμία που θα προκύψει από αυτή τη νέα εταιρική σχέση. Επίσης, ε, για μια τριετία δεσμεύονται όλοι οι μέτοχοι και δεν θα αλλάξει η δομή ε, του μετοχικού κεφαλαίου. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι απόλυτα διαφανή και τα έχουμε δείξει και τα έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη τελευταία διαφάνεια βλέπουμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια τετραετή ε, εταιρική σχέση και αν η αποστολή καθολικής υπηρεσίας του Euronews ή αν οποιαδήποτε αλλαγή στην ιεραρχία και στο μετοχικό κεφάλαιο ε, της Euronews μπορεί η Euronews να αποσυρθεί από αυτήν την τετραετή ε, εταιρική σχέση πλαίσιο. Εάν θέλουμε να στηριζόμαστε από την Ευρώπη, θα πρέπει βεβαίως να κρατήσουμε αυτή την αποστολή παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε για να παρουσιάσω τις θέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν στη με τη συζήτηση, αν θέλουμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καριμπέτη και τον κύριο Αμπαμόντε. Μάλλον έτσι θα το κάνουμε, κύριε Αμπαμόντε. Thanks very much, um, uh, Mrs. Chair. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω. Θα προσπαθήσω να είμαι λιγάκι πιο συνοπτικός από τον προλαλήσαντα. Θα πω δύο λόγια για τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Euronews. Η νομική βάση είναι ε, ο νόμος για τα μέσα και τον προϋπολογισμό και ο στόχος είναι ε, να ενισχύσουμε την ε, παραγωγή νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν είναι μέτοχος του Euronews. η σχέση μας βασίζεται σε ένα, σχέσιο, ε, σε μια, σε ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης όπου αναγνωρίζεται η αποστολή του Euronews για την παραγωγή καθολικής υπηρεσίας. Δηλαδή, ε, θεωρείται μονοπόλιο ε, για την εκπομπή ειδήσεων μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχει και ένας χάρτης αυτή τη συμφωνία για την συντακτική ανεξαρτησία του Euronews. Με βάση αυτή τη συμφωνία, το Euronews θα πρέπει να σέβεται την αρχή της ευρωπαϊκής προοπτικής και της πολυγλωσσίας. Αυτές είναι δύο πολύ σημαντικές αρχές. Δεν θα πρέπει... Είναι σίγουρο ότι οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να παράσχουν το ίδιο περιεχόμενο ούτε σε όλες αυτές τις γλώσσες ε, όπως το Euronews. Γι' αυτό είναι και μαδικό το Euronews η Κομισιόν υπέγραψε μια νέα εταιρική σχέση τετραετή μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Είναι ένα πλαίσιο σύμβασης όπου χάρη στο οποίο η Κομισιόν μπορεί να χρηματοδοτήσει το Euronews σε αιτήσια βάση. Όπως είπε και ο Μάικλ, το πλαίσιο αυτό ε, δεν εγγυάται την πολιετή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να το βλέπουμε το θέμα της χρηματοδότησης ε, χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει. Η Κομισιόν χρηματοδοτεί την παραγωγή και την εκπομπή διαφόρων προγραμμάτων για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ε, σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, αυτά που λέμε μαγκαζίνο ε, οι εκπομπές ειδικέ για την πραγματική οικονομία με ειδικό θεματολόγιο κτλ. για τα ευρωπαϊκά θέματα. Το 2016 η συνεισφορά έφτασε σε 24,8 εκατομμύρια ευρώ, η χρηματοδότηση δηλαδή της Κομισιόν προς το Euronews. Το 2017 η Κομισιόν θα κρατήσει τη χρηματοδότηση περίπου στα ίδια επίπεδα, λίγο πιο χαμηλά, αλλά περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ε, και με βάση αυτό το νόμο ε, για τα ΜΜΕ θα έχουμε και τα φαρσί, τα περσικά. Και επίσης θα χρηματοδοτήσετε ελληνικά, ουγγρικά και πορτογαλικά, καθώς και αραβικά και φαρσί. Θα είναι μόνιμες δηλαδή γλωσσικές αυτές οι εκδοχές. Για τα φάρση λάβαμε ε, μέσα στο 2017, ε, αντί για 3,4 εκατομμύρια το 2016, λάβαμε 3,17 το 2017, λιγάκι, λίγο λιγότερα λεφτά δηλαδή. Λόγω των πρόσφατων αλλαγών στην κεφαλαιοκή δομή του Euronews, το, ε, η συμφωνία του 2017 για τη χρηματοδότηση ε, προβλέπει ότι θα πρέπει να καλύπτει με ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς ε, μεροληπτική παρουσίαση ε, τα νέα, ε, παρέχοντας μία πολύγλωση ευρωπαϊκή προοπτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μηχανισμούς ελεγκτικούς πολύ ισχυρούς, ούτως ώστε το Euronews να σέβεται την Συμφωνία Χρηματοδότησης αλλά να εξασφαλίσει και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, σημαντικό για μένα που είμαι ο διατάκτης, ο χρηματοδοτικός διατάκτης, ότι όλα συμβαίνουν με βάση την αρχή της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει εξωτερική οικονομική έλεγχη που γίνονται σε αιτήσια βάση, καθώς και εξωτερική ανεξάρτητη έλεγχη για αξιολόγηση. Το, η Moore Stevens ε, το 2016 αξιολόγησε την αποτελεσματική σχέση κόστους-οφέλους. Αυτά. Και βρήκε ότι βεβαίως όλες οι δράσεις είναι σύμμορφες προς αυτά που προβλέπονται στη συμφωνία. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι κάνουμε παράλληλους μονολόγους. Έχουμε μια επιστολή των εργαζομένων του Euronews την οποία έχουν υπογράψει όλοι οι εργαζόμενοι, το Επιχειρησιακό Συμβούλιο, το Συνδικάτο του Euronews, όπου ισχυρίζονται ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των περικοπών και των παρεμβάσεων που οδηγούν στον περιορισμό της συντακτικής ελευθερίας, της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι εργαζόμενοι ισχυρίζονται, ε, μάλλον ε, επικρίνουν την απόλυση του Ουκρανικού τμήματος και καταγγέλουν περιορισμούς στο αραβικό και περσικό πρόγραμμα. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα που να απαντά σε αυτές τις καταγγελίες. Ίσως θα μπορούσαμε να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίαση, να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτρες και μετά ξανά στον κύριο Αμπαμόντε, μήπως και μας απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα ε, να πω κάτι εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού. Ως Επιτροπή Πολιτισμού μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε έναν, ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης στην Ευρώπη το οποίο θα ασχολείται κυρίως με ευρωπαϊκά θέματα. Και πέραν του γεγονότος που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι πρώτη φορά που ακούμε καταγγελίες εργαζομένων που ε, αμφισβητούν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του Euronews ως δημοσιογραφικού ε, μέσου. Είμαστε ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού υποχρεωμένοι βεβαίως να τα διερευνήσουμε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε και εμείς δικά μας ερωτήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που δεν μπορούμε παρά να τα, να διερευνήσουμε. Αν δηλαδή το NBC στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας καταλήξει να κατέχει το 85% των μετοχών, δηλαδή βρίσκεται το 85% των μετοχών σε ιδιοκτήτη που έχει την έδρα του εκτός Ευρώπης, μη Ευρωπαίο δηλαδή, ε, δεν μπορεί αυτό να μας αφήσει ε, αδιάφορους ε, όταν, όταν μιλούμε για τον σταθμό εκείνο ο οποίος έχει ως κεντρικό καθήκον του να ενημερώνει τους ευρωπαϊκούς λαούς για τα ευρωπαϊκά θέματα και το να δίνονται 25 εκατομμύρια από τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό στο yes, δεν είναι και αμεληταίο ποσό. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι ε, και εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, το ότι θα μπορούσαν αυτά τα 25 εκατομμύρια να αξιοποιηθούν και πολύ καλύτερα ίσως σε άλλους τομείς. Άρα θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα, ή τουλάχιστον εγώ θέτω αυτό το ερώτημα, ε, Αυτά τα 25 εκατομμύρια τα οποία διατίθενται στο Euronews κάθε χρόνο από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό επιτρέπεται να δίνονται σε έναν ιδιωτικό σταθμό και αν ναι, αυτό πράγματι εξυπηρετεί την ε, αποκόμιση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ιδίως όταν έχουμε διαρκώς καταγγελίες οι οποίες αμφισβητούν την δημοσιογραφική και συντακτική ελευθερία και ανεξαρτησία. Και φαντάζομαι ότι οι εργαζόμενοι του Euronews δεν βλέπουν φαντάσματα, ούτε το έβγαλαν από την κοιλιά τους αυτό. Πιθανότατα ε, να υπάρχει πράγματι κάποιο πρόβλημα σχετικά με αυτά τα θέματα στο Euronews. Και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η σημερινή μα κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να διασκεδάσουμε αν θέλετε αυτέ τι ανησυχίε και αυτέ τι προκλήσει. Και σε αυτό ε, πρέπει, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει βεβαίω να δοθούν απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Γκρέσλε. Τώρα, θα ήθελα να προτείνω να κάνουμε ε, μια συζήτηση ε, να ανοίξουμε τον κατάλογο μολυτών, να τοποθετηθούν τα μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια θα ξαναδώσουμε τον λόγο στον κύριο Αμπαμόντε και τον κύριο Πέτερς για να απαντήσουν. Ο πρώτος ε, στον κατάλογο είναι ο κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τους περιορισμούς για τα Πέρσικα. Ταυτόχρονα υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν και την αραβική γλώσσα, το αραβικό τμήμα. Αλλά εμένα τώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα πέρσικα. Αρχικώς, το μοντέλο χρηματοδότησης ήταν περίπλοκο. Μεγάλο κομμάτι της, ε, του, του, χρηματοδότησης προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τώρα πια ε, τα πέρσικα ε, ακούγεται ότι θα συνεχιστούν στο διαδίκτυο αλλά όχι στην τηλεόραση. Η κατάσταση αυτή είναι σημαντική διότι θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι αφενός το ίντερνετ ε, μπορεί να, τύχει, να, γίνει θύμα ε, Άρα δεν μπορεί κανείς να θεωρεί δεδομένο ότι όλες οι ειδήσει φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους Αλλά ακόμη χειρότερα, ε, είναι πλέον ε, τεχνολογικά δεδομένο ότι ε, μπορεί κανείς να παρακολουθεί ε, τους ανθρώπους εκείνους μέσω του διαδικτύου που, εκεί, που παρακολουθούν ειδήσει που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Δυστυχώς υπάρχει. Υπάρχουν λογισμικά που μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν τέτοιο σκοπό. Γι' αυτό για τους ανθρώπους που ζουν στο Ιράν είναι, επικίνδυνο να παρακολουθούν Euronews στα περσικά. Εκτός Ιράν φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, αυξάνεται και ραγδαία ο αριθμός των χρηστών. Αλλά η διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού προγράμματος, που είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί από την κυβέρνηση του Ιράν, θεωρώ ότι είναι καταστροφή. Είναι, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την εξωτερική μας πολιτική και θα αποδυναμώσει τις δυνάμεις με τις οποίες θέλουμε εμείς να συνεργαστούμε στο Ιράν βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας για 700.000 ευρώ. Αξίζει πραγματικά. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω. Ευχαριστώ πολύ Ραμπέκα Χάνς. Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική αιτιολόγηση λόγω των πολιτικών, των πολιτικών εντάσεων που έχουμε γύρω από το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν μπορεί να δοθεί για τη διακοπή του Ουκρανικού, του Τουρκικού και του Περσικού προγράμματος. Αντιθέτως, η απάντηση θα έπρεπε να είναι ότι αυτά τα τρία προγράμματα πρέπει να συνεχιστούν πάση θυσία και με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε αυτές τις εταιρικές αποφάσεις του Euronews ελπίζω οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται μόνο με, με όρους ιδιωτικής οικονομίας και ανταγωνισμού, αλλά ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Επίσης θα με ενδιέφερε πώς μπορούν να συνδυαστούν οι δραστηριότητε του Euronews με τις δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας. Σε πολλές επιτροπές έχουμε συζητήσει για, το, για την μάχη της προπαγάνδα προπαγάνδας που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο τι σημαίνει ε, για την, ανεξαρτησία του Euronews όταν υπάρχουν Ρώσοι χρηματοδότες του Euronews και αυτό οδηγεί στο να διακόπτεται η λειτουργία του, του Ουκρανικού προγράμματος και οδηγεί επίσης στη συνέχιση του Ρωσικού προγράμματος. Συγκεκριμένα για το Ουκρανικό πρόγραμμα. Άκουσα ότι οι δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Ουκρανικό ε, πρόγραμμα προσπαθούν να συνεχίσουν τη λειτουργία αλλά το ότι δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουν τη δουλειά τους λόγω του γεγονότος ότι είναι Ουκρανοί πολίτες. Η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας παρατρύνω κυρία Γκρέσλε να σχολιάσετε την επιστολή που λάβαμε διότι διαβάζοντα την καθίσταται σαφέ ότι αντιμετωπίζει κρίση, κρίση η Euronews και δεν το αναφέρατε. Ε, είναι προφανής η κρίση αυτή και έτσι θα ήθελα να μου πείτε σε ποια έκταση οι επικρίσεις που ακούμε από το προσωπικό της Euronew's σχετίζονται με τα εμπορικά ζητήματα. Εσείς είπατε ότι ο αντιγωνισμός είναι υψηλός και ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όσον αφορά τα διάφορα επιχειρηματικά ζητήματα το Μέσο μαζικής ενημέρωση παγκοσμίω. Ήθελα λοιπόν να επανέλθω στο γενικότερο ερώτημα οφείλεται στο ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις πολιτικές μας φιλοδοξίες για ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ειδήσει ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερω να έχουμε ε, δημόσιες ειδήσει ε, που να καλύπτουν τις ειδήσει όπως επιθυμούμε εμείς και ακούγοντάς σας είναι σαν να μου λέτε ότι δεν είστε πλέον σε θέση για κάτι τέτοιο. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι με όλη αυτή τη δομή, με τι εμπορικέ δεσμεύσει, με την εξέβρεση νέων επενδυτών. Θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι πολιτικοί μα στόχοι. Αν δει κανεί την πολιτική γειτονία ε, και το τι κάνει η Γερονιό, δεν υπάρχει αντιστοιχεία αυτών με το τι κάνουμε εμεί τι πολιτικέ γειτονία. Οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι, χρειαζόμαστε μια πραγματική μήπω δημόσια δομή τη Euronews, ώστε να μπορούμε να ε, κοινοποιούμε ε, τους πολιτικούς μας στόχους ε, και να τους επιτυγχάνουμε. Αυτή είναι ε, η ερώτησή μου και στο μέλλον η ερώτησή μου θα είναι ποια θα μπορούσε να είναι μια ασφαλής βάση για τη Euronews γιατί ακούγοντάς σας δεν αποκόμισε την εντύπωση ότι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή διασφαλίζει το μέλλον της Euronews ούτε τις πολιτικές φιλοδοξίες που επιδιώκουμε εμείς μαζί με τη Euronews. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Άλλος ένας ομιλητής βρίσκεται στο κατάλογο μολυτών και μετά θα ε, δώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτερς και τον κύριο Αμπαμόντε. Λουίτζι Μοργκάνο. Ευχαριστώ. Είναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε εδώ λόγω του προβλήματος που υπάρχει. Έχουν γίνει και στο παρελθόν συζητήσεις. Εγώ θα ήθελα να σας απευθύνω τέσσερις ερωτήσεις μου φαίνονται σημαντικές. Ακούσαμε μεγάλη σαφήνεια ότι η συμφωνία είναι τετραετής, έτσι όχι τριετής, μου λέτε. Και κάθε χρόνο επαληθεύονται εκ νέου οι οικονομικές συνθήκες. Και υπάρχει έλεγχος ε, της σύνταξης από το δημόσιο μέτοχο, έτσι, από το δημόσιο δηλαδή. Και ο έλεγχος του προπολογισμού γίνεται ε, και ο δημόσιος μέτοχος έχει το 85% του προϋπολογισμού. Λοιπόν, συγκεκριμένα ερωτήματα. Σε αυτά τα 25 χρόνια που υπάρχει το Euronews, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι φορέα έχει δημιουργήσει για να στηρίξει το Euronews. Μας μιλήσατε για την ανεξαρτησία, μας μιλήσατε για τους πολιτικούς στόχους, μας είπατε ότι τα προγράμματα παρουσιάζουν σωστά την πραγματικότητα. Όμως, το σχέδιο για τη σύνταξη, το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή κερδίζουμε τέσσερα χρόνια, αλλά για να προωθήσουμε κάτι το οποίο είναι εντελώ άμορφο ακόμα. Επίσης, η παραχώρηση του Eurosport του Eurosport αξιολογήθηκε το 2015 σε ένα δισεκατομμύριο. Έτσι. Με, με αυτό το δεδομένο θα ήθελα να καταλάβω το συνολικό πλαίσιο που έχουμε. Euronews, Eurosport κτλ. Ευχαριστώ Λουίτζι. Κύριε Πέτερς, έχετε το λόγο. Um, thank you very much. I would just like to thank you, Mrs. Camerabert, to have um, Ευχαριστώ τη συνάδελφο που έθεσε το σωστό πλαίσιο για τη συζήτηση σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και γι' αυτό ήρθα εδώ, για να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις και να προσπαθήσω να σας πείσω ότι κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει, σωστά. Καλό είναι το να υπάρχουν ερωτήσεις, αλλά είναι άλλο το να κατηγορεί κανείς. Είναι κάτι που δεν θα δεχτώ. Και θα λάβουμε όλα τα μέτρα εναντίον των ανθρώπων που μας κατηγορούν. Μάλιστα, άκουσα διάφορες ερωτήσεις. Καταρχάς για τις γλώσσες. Τα φάρση, τα ουκρανικά και τα αραβικά. Καταρχάς, να σας εξηγήσω Είμαι εδώ σαν επιχειρηματίας, έτσι, όχι σαν πολιτικό. Προσπαθώ να διευθύνω μία ιδιωτική εταιρεία. Ακόμα και όταν το 100% των μετοχών τα είχε το δημόσιο, ήταν ανεξάρτητη. Και έχουμε και συμβάσεις ούτως ή άλλως. Παλιά είχαμε συμβάσεις με την Εθνική Τηλεόραση της Ουκρανίας. Ε, πρέπει να σας πω ότι η Ουκρανική Εθνική Τηλεόραση μας ε, χρωστάει 10 εκατομμύρια. Τα τελευταία, δηλαδή, δύο χρόνια δεν μας πλήρωσε και έχουμε πάει στα δικαστήρια για να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Δεν έχουμε κάποιον εταίρο αυτή τη στιγμή που θα μπορέσει να ε, χρηματοδοτήσει αυτές τις γλώσσες. Δεν είμαστε εμείς από την άλλη σε θέση οικονομική. Βεβαίω άκουσα από εσά επιχειρήματα πολιτικά, ε, συντακτικά. Ε, το θέμα είναι οικονομικό. Εγώ δεν είμαι σε θέση να ζητήσω από τους μετόχους ούτε το, το δημόσιο, αλλά ούτε και τους ιδιωτικούς μετόχους να χρηματοδοτούν αυτές τις γλώσσες που δεν αποφέρουν έσοδα τη στιγμή που η εταιρεία χάνει λεφτά. Η απόφαση να σταματήσουμε την εκπομπή στα Ουκρανικά δεν ήταν πολιτική απόφαση, δεν ήταν απόφαση τη ε, σύνταξη. Ήταν μια οικονομική απόφαση. Δεν έχουμε τα μέσα να χρηματοδοτήσουμε ή μάλλον να αυτοχρηματοδοτηθεί μια γλώσσα. Είναι μια οικονομική πραγματικότητα, έτσι και το υπογραμμίζω. Εγώ είμαι αυτός που ξεκίνησε τις εκπομπές στα Ουκρανικά. Καταλαβαίνω τη σημασία την πολιτική σημασία των εκπομπών στα Ουκρανικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τα οικονομικά μέσα να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε στα Ουκρανικά. Για τα Ρωσικά τώρα. Άκουσα ένα λάθος ε, επιχείρημα. Η ρωσική γλώσσα, η εκπομπή στα ρωσικά, δεν χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος. Είναι λάθος. Όπω είπα και στην παρουσίαση, τα ρωσικά αυτοχρηματοδοτούνται από το Euronews. Πώ γίνεται, γιατί η ρωσική γλώσσα είναι σήμερα το 35% του συνολικού ακροατηρίου του Euronews. Είναι τεράστιο νούμερο. Γιατί είμαστε ίσως ε, το μόνο εξάρτητο μέτρο, μέσο το οποίο δεν βασιζόμαστε στη, στο ρωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο για, τα, για τις ειδήσει μας. Αν χάσουμε τη ρωσική γλώσσα στο Euronews θα χάσουμε 30 με 35% του ακροατηρίου μας, των θεατών μας. Και αυτό θα είναι οικονομική καταστροφή για την εταιρεία. Και μάλιστα, χάρη στα ρωσικά, έχουμε ένα εργαλείο έκφρασης, ευρωπαϊκό εργαλείο, που χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Ρωσία και το ρωσικό κοινό. Αυτά λοιπόν για τη ρωσική γλώσσα. Τώρα, για το τι θα, απογίνει το ουκρανικό προσωπικό. Τι θα γίνουν αυτοί οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι. Άκουσα κάποια λάθος πράγματα. Προσπαθούμε να τους βάλουμε σε άλλα πόστα. Και μάλιστα θα πούμε σύντομα στο προσωπικό ότι κάποιοι, λίγοι από αυτούς, θα πάνε σε άλλα τμήματα του Euronews, σε άλλες θέσεις. Τώρα, για, το, για τα φάρση. δεν είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι απόφαση τη σύνταξη. Το ξαναλέω, έχουμε μια εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την, ε, την Υπηρεσία εξωτερική δράση της ε, κυρίας Μογκερίνη, η οποία αποφάσισε να μειώσει κατά πολύ τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός ήταν, ήταν 5 εκατομμύρια, έγινε 4 και μετά 3. Σωστό. Από 5 πήγε 3 δηλαδή. Και με αυτό το προϋπολογισμό δεν μπορούμε να προσφέρουμε μία επαγγελματικά σωστή ε, εκδοχή, ας πούμε, στα φάρση. Επομένως, θα, δει θα εκδίδεται το περιεχόμενο αυτό στα φάρση μόνο μέσω ίντερνετ. Ψηφιακά δηλαδή. Φυσικά, αν αυξηθεί ο προπολογισμό, θα ξαναβάλουμε, θα ξανανεβάσουμε τα φάρση στην τηλεόραση. Προσπαθώ να βρω έναν άλλο εταίρο, ούτω ώστε να ξαναβάλουμε τα φάση στην τηλεόραση. Αλλά στο ψηφιακό κομμάτι είναι περίεργο. Αλλά η περσινή εκπομπή έγινε η τρίτη πιο σημαντική εκπομπή στο ίντερνετ. Σε φάση, έτσι. Η εκπομπή δηλαδή του Euronews. Και το Ιράν είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο που καταναλώνει το Euronews. Δηλαδή η τρίτη μεγαλύτερη. Χάρη σε αυτές τις νέες τεχνολογίες μπορούμε σήμερα να παρακάμψουμε τα διάφορα φίλτρα που μπαίνουν. Και πρέπει να σας πω ότι τα φάρση λειτουργούν άψογα σε ψηφιακό υπόθεμα. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι με το στρατηγικό διάλογο που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθούμε ένα στόχο κοινό, έτσι, να περάσουμε ε, και να μετα... εκπέμψουμε περισσότερο στο ίντερνετ σε ψηφιακό υπόθεμα. Ε, ειδικά για αυτές τις γλώσσες, φαρσί, αραβικά. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ε, ψηφιακή στρατηγική για αυτές τις γλώσσες. Και πριν πω στο βασικό θέμα, θέλω να πω κάτι για το Eurosport. Το ρώτησε η κυρία Τσούπελ. Δεν μπορώ να σχολιάσω για αυτό το ένα δισεκατομμύριο ε, η αξία της εκχώρησης λίστα του Eurosport. Ξέρετε ότι υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα. Από αυτό αποτελείται το Eurosport. Δεν ισχύει αυτό για το Euronews, δυστυχώς. Εξού και το ύψος αυτό του ποσού, το μεγάλο ποσό αυτό. Πάντως, ε, φυσικά ο στόχος των διευθυντών του Euronews είναι να ανεβάσουμε την αξία μας τα, τα επόμενα χρόνια. Τώρα μπαίνω στο ψητό. Καταλαβαίνω απόλυτα το ότι ανησυχήσατε, θορυβηθήκατε από αυτή την επιστολή που έγραψε το προσωπικό. Ναι, όντως, σωστό. Υπήρξε μια κοινωνική κρίση τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω του ότι καταρχάς σταματήσαμε να εκπέμπουμε στα Ουκρανικά, που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είχαμε, μας οδήγησε σε περικοπές ε, θέσεων απασχόλησης στο Euronews και φυσικά αυτό κοινωνικός πως φυσικά δεν δημιουργεί, δεν είναι καλό και το κλίμα σίγουρα επιδεινώνεται προφανώς. Επίσης, ε, τα αραβικά και τα φάρση εκπέμπονται πια μόνο ε, στο ίντερνετ, σε ψηφιακό υπόθεμα. Φυσικά, οι σχετικές ομάδες ε, δυσαρεστήθηκαν. Θα προτιμούσαν να συνεχίσουν να δουλεύουν στην τηλεόραση, αντί για το ίντερνετ. Αλλά πέραν τούτου, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά στο Euronews από τον κόσμο και από τις ομάδες που ήρθαν στο Euronews πριν από 25 χρόνια για να δουλέψουν σε ένα καθαρό δημόσιο οργανισμό. Γιατί το Euronews χρηματοδοτούνταν 100% από το δημόσιο τότε. Και οι περισσότεροι ε, που δουλεύουν στο Euronews δουλεύουν και 20 χρόνια. Και το γεγονός ότι το Euronews στρέφεται σε πιο εμπορικά σχήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν κολλάει με την αντίληψη που είχαν ε, αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν στο Euronews. Το θέμα είναι, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό λοιπόν. Δεν έχω την απάντηση. Βοηθήστε με. Αυτό που έχω είναι το δημόσιο που δεν θέλει πια να χρηματοδοτεί το Euronews. Αυτή είναι η κατάσταση. Αφού δεν θέλει να μας χρηματοδοτεί πια, εμείς θα πρέπει να στραφούμε σε ιδιωτικούς επενδυτές. Αυτή η επιστολή επίσης γράφτηκε και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Είναι σημαντικό να καταλάβετε πότε γράφτηκε αυτή η επιστολή. Γράφτηκε όταν περιμέναμε να υπογραφεί η Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία υποτίθεται θα υπογραφόταν τον Οκτώβριο, μετά αναβλήθηκε για το Δεκέμβριο και μετά για τον Ιανουάριο, αναβλήθηκε, λογικό, θεμητό, λόγω των συζητήσεων που έγιναν και που γινόταν με το NBC. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε δεν μπορούμε να υπογράψουμε την συμφωνία πλαίσιο χωρίς να ξέρουμε θα συμβεί με το NBC. Και πώς το Euronews θα βάλει τις ασφαλιστικές δικλείδες ούτω ώστε να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της σύνταξης. Ανησυχούσαμε λοιπόν στο Euronews, όλο το προσωπικό ανησυχούσε, ε, γιατί φοβόταν πως δεν υπογραφεί καν αυτή η συμφωνία πλαίσιο. Ο χρονισμός ήταν πάρα πολύ σημαντικός, γιατί τη στιγμή που υπογράφηκε αυτή η επιστολή από το προσωπικό, το ξέρω πολύ καλά, εμείς θέλαμε να ζητήσουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ζητήσουμε αυτή η πολιετή συμφωνία πλαίσεων να υπογραφεί. Αν θέλετε ξαναδιαβάζουμε την επιστολή. Την ξαναβλέπουμε μαζί με οποιονδήποτε θα το ήθελε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος για την ανεξαρτησία μας. Α, την ανεξαρτησία μας απέναντι στους ιδιωτικούς ε, επενδυτές. Θα σας πω κάτι. Το Συμβούλιο ε, της Επιχείρησης του ε, Euronews που εκπροσωπεί όλους τους εργαζομένους και όλους τους, όλα τα συνδικάτα ομόφωνα ε, υπερψήφισαν το MSNBC. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη από αυτή που έχει εμφανιστεί. Ε, βεβαίως ε, προσπαθούμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις των εργαζομένων. Υπάρχει θλίψη και δυσαρέσκεια Υπάρχουν βεβαίως κάποιοι ε, συνάδελφοι οι οποίοι θα ε, είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουν, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει, αν θέλουμε να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε, να αλλάξουμε. Αν δείτε και τι γίνεται στο ευρύτερο πλαίσιο. Και να τελειώσω με το ερώτημα, από ό,τι κατάλαβα, που είναι στην ουσία αν σε τελική ανάλυση το Euronews θα πρέπει να είναι δημόσιος οργανισμός ε, που θα εξυπηρετεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ πιστεύω όχι. Η απάντηση κατά την γνώμη είναι όχι. Το ερώτημα δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώ και του ε, μετόχους. Το ερώτημα είναι τι θα προσφέρει στους καταναλωτές της Ευρώπης το Euronews. Και αυτό που πιστεύω ακράδαντα και ίσως δεν καταφέρω να σας πείσω είναι ότι το σχέδιο που έχουμε με το ε, MSNBC δεν είναι πολιτικό σχέδιο. Είναι ένα business plan, ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν έχουν... Ε, ε, δεν έχουν αυτή τη στιγμή ε, θέση ε, πλην του Euronews στην, στην Ευρώπη. Το, το Euronews είναι το πλέον δημοφιλές μέσο ευρωπαϊκών ειδήσεων. δεν μπορείς όμως να επηρεάζει τα πράγματα. αν θέλεις να μιλήσεις για, τα, για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και να αλλάζεις τις γνώμες των ανθρώπων, χρειάζεσαι και τα κατάλληλα μέσα, τα format, ε, talk show, συνεντεύξεις, μεγάλα show, το οποίο θα σου, δώσουν, θα σου τη δυνατότητα να έχεις ε, κόσμο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και από τους δρόμους ε, απλούς Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι θα βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να σχηματίσουν τη δική τους γνώμη. Αυτό είναι και το πρόγραμμα, το σχέδιο που έχουμε με το MSNBC. Το MSNBC θέλει να επενδύσει πολλά χρήματα προκειμένου να μπορέσει να προτείνει νέα φορμάτ, τα οποία θα μας βοηθήσουν να διανύμουμε το δικό μας ε, περιεχόμενο. Θέλουμε να κάνουμε δημοσιογραφία βάσης σε αυτό θα μας βοηθήσει η συνεργασία με το MSNBC. Θα δώσουμε λόγο στους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά αφορούν τα επιχειρηματικά σχέδια. Και πρέπει να σας πω ότι δεν βρέθηκε κανένας άλλος εταίρος που να ενδιαφέρεται κάτι τέτοιο και κανένας άλλος Ευρωπαίος εταίρος. Εγώ συζήτησα με 80 διαφορετικά δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Μίλησα με δημοσιογραφικούς ομίλους από τη Γερμανία, από τη Γαλλία. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για το ε, Euronews. Και το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους εκτός Ευρώπης οι οποίοι θέλουν να μας βοηθήσουν να, να καταστήσουμε το Euronews ε, πιο αποτελεσματικό και να αυξήσουμε την, ε, την επιρροή του. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Γκαριμπέρτη, θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο ανοιχτά να εκφράζονται εδώ μέσα απειλές κατά εκείνων που έχουν απευθυνθεί σε εμάς Ω Επιτροπή Πολιτισμού και Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού με τι ανησυχίε του. Το κάνατε αυτό στην αρχή τη ομιλία σα, στην πρώτη σα τοποθέτηση. Παρακαλώ ανακαλέστε ή διορθώστε. Σω καταλάβαμε κι εμεί λάθο την τοποθέτησή σα, αλλά πρέπει να σα πω ότι ε, εγώ εξέλαβα αυτά που είπατε ω απειλή. Και νομίζω ότι σε μια τέτοια αίθουσα κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και σε δημόσιο χώρο, αλλά και κεκλεισμένων των θυρών να συνεδριάζαμε. Πάλι απαράδεκτο θα ήταν. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκαριμπέρτη. Mm, Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα. Η επιστολή στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως μου θυμίζει ε, τότε που ψηφίστηκε χρεοκοπία της Αλιτάλια για να μην γίνει δεκτό ένα σχέδιο το οποίο θα περικοπτε, ε, περικοπτε πολλές θέσεις εργασίας. Είναι σαν τον ε, ε, σκορπιό που μεταφέρεται στην άλλη οχθή του ποταμού από ένα βάτραχο και μετά τσιμπάει το βάτραχο. Εγώ όταν έγινα πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Euronews το 2012, όταν τελείωσα ε, ως πρόεδρος της ΡΑΕ ε, και εγώ ξέρετε είμαι δημοσιογράφος ε, και στον τύπο και στην τηλεόραση. Όταν έγινα λοιπόν πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Euronews, Euronews ήταν πράγματι μια επιχείρηση τηλεοπτική δημόσια από όλες τις απόψεις, διότι χρηματοδοτεί το μόνο από τους δημόσιους ε, ε, μετόχους. Τότε η ΡΑΗ έδωνε 1,4 εκατομμύρια ευρώ, η γαλλική ε, τηλεόραση το ίδιο και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή οι δημόσιοι μέτοχοι ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να μειώσουν σταδιακά τις χρηματοδοτήσεις τους μέχρι να τις μηδενίσουν από το 1,4 στο 0. Οπότε κατέστη απαραίτητο γιατί να επιβιώσει η Euronews να βρει άλλους εταίρους. Ούτως και πράξαμε μετά από δύο χρόνια έρευνας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Πέτερς, το πράξαμε με την τελική συνένεση της Κομισιόν, με την οποία διαπραγματευτήκαμε για πολύ καιρό την εισαγωγή ενός ε, ε, ιδιωτικού ε, επενδυτή ώστε να επιβιώνει η Euronews. Διαφορετικά θα χανόταν. Όσοι λένε λοιπόν θα θέλαμε να μείνουν τα πράγματα όπως πριν από 25 χρόνια όταν ιδρύθηκε η Euronews πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει και ότι η Euronews θα χαθεί αν δεν χρηματοδοτηθεί από αλλού. Αυτά όσον αφορά ε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Από τότε που μπήκε ο Ναγκή Ψαβήρης και εγώ έγινα πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και του Συντακτικού Συμβουλίου με την αρμοδιότητα να επαληθεύω κατά πόσο ο News διατηρεί ε, τις διασφαλίσεις ανεξ, ε, ανεξαρτησίας που ε, την είχαν χαρακτηρίσει όλα αυτά τα χρόνια με τους δημόσιους μετόχους μπορώ να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτή την άποψη. Η ποιότητα μάλιστα της Euronews έμεινε άθικτη και η αποτελεσματικότητα της Euronews όσον αφορά τη διαβίβαση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών αξιών έχει μάλιστα βελτιωθεί. Πριν από λίγο κάποιος μίλησε για έναν υβριδικό πόλεμο που ε, συντελείται στην Ευρώπη. Εγώ συμφωνώ. Έγραψα και ένα άρθρο σύμφων, ε, πρόσφατα και αυτό ο υβριδικό πόλεμο προέρχεται από κάποια τηλεοπτικά κανάλια, αυτά που χρηματοδοτούνται από τη Ρωσία κυρίω, τα οποία διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο. Ε, η Sputnik, η Russia Today, διάφορα τέτοια κανάλια τηλεοπτικά ή στο διαδίκτυο διαδίδουν ε, τα πιστεύω του Κρεμλίνου. Όταν έγινε η διαδήλωση κατά του Πούτιν, που ε, κόπηκε στο διαδικτύο στη Μόσχα. Ποιος μίλησε για αυτή τη διαδήλωση ενώ την λογόκριναν ε, τα ρωσικά μέσα η Euronews την παρουσίασε. Καμία, κανένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Η CNN Τουρκίας, ε, αντιθέτως, όταν έγιναν διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν, στο τουρκικό κομμάτι της CNN μίλαγε, είχε ένα ντοκιματέρ για τους πιγκουίνους και μάλιστα τη χαρακτήρισαν Penguin Television. Ε, δεν μεταδόθηκε τίποτα στα τουρκικά. Αν σταματήσει η Euronews στα τουρκικά, θα, αυτό θα, τις ευθύνες θα πρέπει να τις ζητήσετε από τον Ερντογάν. Αυτό θα το έχει απαιτήσει. Διότι η τουρκική τηλεόραση, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι κατά του Ερντογάν. 100%. Ο Ερντογάν το αποφάσισε αυτό. Και εγώ σας το λέω ως δημοσιογράφος και αυτή είναι η άποψή μου. Και πιστεύω ότι η άποψή μου θα πρέπει να την υπολογίσετε. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, μέχρι στιγμής δεν είχε αλλάξει τίποτα όσον αφορά την συντακτική ανεξαρτησία της Euronews. Μάλιστα πρόσφατα, περίπου ένα-δύο χρόνια, ε, ε, πριν από ένα-δύο χρόνια, κατηγορήθηκε η ρωσική υπηρεσία της Euronews ότι ευνοούσε υπερβολικά την πολιτική γραμμή του Κρεμλίνου. Κάναμε μια ανεξάρτητη έρευνα που αναθέσαμε ε, στον ε, οργανισμό ελέγχου Παδία ε, ο οποίος εξέτασε κατά πόσο υπήρχε πολιτική ισορροπία της γενικής ενημέρωσης και ο οποίος συνέταξε μια έκθεση στην οποία δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή που να λέει ότι ε, η ρωσική Euronews υποστηρίζει τη γραμμή του Κρεμλίνου. Σε καμία περίπτωση. Και τότε μενόταν η μεγάλη κρίση με το Κρεμλίνο, με την Κρυμαία, συγγνώμη. Ε, και έτσι λοιπόν εγώ ως πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής μπορώ να σας πω ότι οι ιστορίες ε, δίθεν μη ανεξαρτησίας της Euronews είναι ψεύδι. Είναι μύθι. αν πρόκειται να μειωθεί η ανεξαρτησία της Euronews, εγώ θα απαραίτημουν αμέσω. Η καλή δημοσιογραφία, κύριοι, λοιπόν, δεν γίνεται βάση ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Γίνεται διότι ε, κάποιος είναι καλός δημοσιογράφος. Οπότε η καλή δημοσιογραφία πρέπει να διασφαλίζεται από του ίδιου δημοσιογράφου. Αλλά η νοοτροπία τη δημόσια υπηρεσία που γνώρισα εγώ και στη ΡΑΕ είναι ότι καθιστά γραφειοκρατική δημοσιογραφία. Κάτι πολύ εύκολο. Παίρνει κανεί το μισθό του και συμπληρώνει ειδήσει. Αν θέλει να διατηρήσει κανεί την ανταγωνιστικότητα και σε πολιτικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτού του ευρωδικού πολέμου στην Ευρώπη, πρέπει κανεί να κάνει σωστή δημοσιογραφία και όχι γραφειοκρατική δημοσιογραφία. Σε αυτό συνίσταται όλο το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ευχαριστώ. Πρέπει να επιβεβαιώσω και να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κύριος Γκαριμπέρτη και με όσα είπε ο κύριος Πίτερς. Πρώτον, σχετικά με το παρατηρητήριο της Παβία, το οποίο είναι ε, μια οντότητα με μεγάλο κύρος. Σκοπός του Euronews uh, uh, um, είναι να αντικρούσει τις ε, κατηγορίες και τους κινδύνους ε, εξαγοράς του. Υπήρξε πράγματι μια καταγγελία ε, μεροληψίας υπέρ του Κρεμλίνου στην ειδησογραφία του Euronews. Το παρατηρητήριο εξέτασε και διερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε στο ότι η κατηγορία αυτή ήταν αβάσιμη. Μάλιστα προέβη σε μια σειρά από αξιολογήσεις για το Euronews. Υπήρξε, για παράδειγμα, ε, ε, έλεγχος λογιστικός το 2016, η Lloyd έκανε κάτι παρόμοιο το 2014 και βεβαίως ανέκυψαν κάποια ζητήματα. Δύο συγκεκριμένα. Πρώτον, ήταν η μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική βιωσιμότητα του μοντέλου του Euronews και η κίνδυνοι που προκύπτουν από τη μείωση της χρηματοδότησης των κρατικών ε, σταθμών. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν ότι το, μοντέλο του, το επιχειρηματικό μοντέλο του Euronews, όπως και άλλων οργανισμών δισογραφικών, θα πρέπει να προσαρμοστεί στην νέα ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθούν νέες ε, δυνατότητες, ε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει ε, ούτε ο λογιστικός έλεγχος την ανεξαρτησία της σύνταξης του Euronews. Εξ όσων γνωρίζουμε λοιπόν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την ανεξαρτησία αλλά και την ευρωπαϊκή γραμμή την οποία υπηρετεί το Euronews και σε αυτή, αυτό είναι που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο για, ε, για, τα, για το πρόγραμμα ε, στην περσική γλώσσα είπατε ότι ξοδεύουμε πολλά χρήματα για το Euronews. Ε, δεν είναι και πολλά, διότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για παράδειγμα, το, το τρέχον, το 2014-2020 για τις ε, δράσεις πολυμέσων ε, προέβλεπε 20% μείωση. Κατά συνέπεια, αυτό είναι, αυτή είναι, αυτό είναι το οικονομικό περιβάλλον. Ο, οι προπολογισμοί περικόπτονται και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να αξιοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το ίδιο αφορά και τη χρηματοδότηση από την ΕΕΔ. Το είπε και ο Μάικλ Πίτερς ότι ε, μας είπε η Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι ε, μειώθηκε η χρηματοδότηση και έτσι ήταν ε, αναγκαίο να περιοριστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο διαδίκτυο και μόνο. Και μάλιστα από ό,τι μας είπε και ο Μάικλ η επιλογή αυτή στέθηκε με επιτυχία. Και τέλος, Υπάρχει και ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο. Για το NBC η συμφωνία δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ οι διάφορες λεπτομέρειες της συμφωνίας ε, βρίσκονται ακόμη υποσυζήτηση, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Θα συνεχίσουμε να, να, να παρακολουθούμε το ζήτημα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση, με τον κύριο Πίτερς και τον κύριο Γκαριμπέρτη και αν αλλάξει κάτι φυσικά θα, αναπροσαρμόσουμε και εμείς τη στάση μας. Αλλά ε, επί του παρόντος δεν έχουμε λόγους να, να αμφιβάλλουμε ε, ε, ή να έχουμε ανησυχίες ότι η συμφωνία με το NBC θα ε, επηρεάσει ε, την, ε, την ποιότητα του Euronews. Αντιθέτως έχουμε την εικόνα ότι θα βελτιωθεί και η, η βιωσιμότητα, η χρηματοδοτική βιωσιμότητα αλλά και η ποιότητα του περιεχομένου που προσφέρει το Euronews. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαμόντε. Έχω δύο ευρωβουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε σύντομα όμως, προκειμένου να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε το λόγο στους κυρίους Πέτερς και Αμπαμόντε. Γιατί στις 4.30 θα πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. να τόν. Ε, έχω τρει ε, σελίδε ερωτήσεων και εσεί μου λέτε να είμαι σύντομη. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Είμαι πρώην δημοσιογράφο και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κύριο Πίτερ. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι κάνουμε λάθος όταν ε, μιλάμε για το Euronews. Λες και είναι μια κλασική, ένας κλασικός φορέας. Αν θέλουμε να είναι θα πρέπει να αφήσουμε τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουμε το Euronews όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται. Από ίδια εμπειρία ξέρω ότι τα κρατικά μέσα, ιδιοσιογραφικά ας πούμε, είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Αφήστε με να τελειώσω. Στην πραγματικότητα κολακεύουν το κοινό. Ε, δεν το βάζουν να σκεφτεί πάνω στα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτή η ισορροπία. Αλλιώ ποτέ θα τα καταφέρει κανένα μέσο ενημέρωση. Έχω και μια έντονη ερώτηση. Στη σελίδα 3 και συγγνώμη που καθυστέρησα. Ίσως το συζητήσατε. Υπάρχει μια διαφάνεια που μιλάει για την αποτελεσματικότητα. Πώς τη μετράτε. Στην πρώτη διαφάνεια της σελίδας 3 λέτε ότι έχετε τεράστιο κοινό. Ε, για την τηλεόραση, έτσι, και στις επόμενες δύο διαφάνειες δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Πώς συγκρε... συγκρίνεται, ας πούμε, την ε, σχέση κόστους-οφέλους με τα άλλα κανάλια. Πιστεύω ότι είσαστε πολύ πιο ακριβοί. Πιστεύω από τους άλλους. Σωστό ή λάθος. Και αν ναι, γιατί είστε πιο ακριβή, παρακαλώ. Ευχαριστώ Γιάννα για το ότι μας τα και τόσο σύντομα. Κύριε Μπούχμαν, πολύ σύντομα θα σας πω κι εγώ. Θέλω να ρωτήσω, οι περικοπές στις γλώσσες φάρση, στο τηλεπτικό, στα αραβικά και στα ουκρανικά στην ουσία οφείλονται στα περιορισμένα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Για το ερώτημά μου προς τις δύο επιτροπές που συνεδριάζουν. Πόσο σημαντικό είναι για εμάς ε, ε σημαντικές είναι, πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση που πηγάζει, που προέρχεται από την, ε, από την Ευρώπη. Δεν είναι και αυτό ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής για να χτίσουμε γέφυρες με χώρες που περνούν δύσκολες εποχές. Μιλώ για την Ουκρανία και το, και το Ιράν. Νομίζω ότι εδώ η εξωτερική πολιτική δράση θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι αξίζει αυτά τα λίγα ευρώ. Και επαναλαμβάνω, 700.000 ε, ευρώ είναι όλο και όλο το κόστος του τηλεοπτικού προγράμματος στα περσικά. Το ερώτημά μου είναι και, και η έκκλησή μου προς τις δύο επιτροπές είναι δραστηριοποιηθείτε γιατί είναι σημαντικό ε, για την Ευρώπη. Η κυρία Γκρέσλε, δύο ερωτήματα. Το ένα για τον κύριο Πέτερς. Η οικονομική βάση των αποφάσεών σας αμφισβητείται με το επιχείρημα ότι στην πραγματικότητα έχετε λάβει μια πολιτική απόφαση. Μήπως θα μπορούσατε να, να μας παρουσιάσετε ποιες ήταν οι άλλες εναλλακτικές σας ε, ε, αποφάσεις και τις οποίες δεν προκρίνατε. Υπάρχουν διάφορες γλώσσες, γερμανικά, ιταλικά κτλ. κτλ. Για ποιο λόγο οι επιχειρηματικές σας αποφάσεις ε, αφορούν τελικά αυτές τις τρεις γλώσσες, ουκρανικά, αραβικά και φαρσί. Μήπως, θα, ε, μήπως υπήρχε δυνατότητα να, ληφθού, να ληφθεί μια διαφορετική αποφάση. Ο κύριος ε, Αμπαμόντε είπε ότι ο λογιστικός έλεγχος δεν κατέδειξε στοιχεία για την ε, ε έλλειψη ε, ανεξαρτησίας του Euronews. Ήταν πραγματικά αυτό αντικείμενο του λογιστικού ελέγχου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να ξαναδώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πέτρες και τον κύριο Αμπαμόντε και να τους παρακαλέσω να μην υπερβούν τα τρία λεπτά. Κοιτάξτε λίγο και το ε, ρολόι σας, ώστε να έχετε περίπου μια εικόνα για το πόσο έχετε μιλήσει. Κύριε Πέτερς. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Η σχέση κόστος ωφέλους στους τελευταίους δύο οικονομικούς ελέγχους ε, διαπιστώθηκε ότι η Euronews ε, είναι η πιο οικονομικά αποδοτική οργάνωση ειδήσεων στην Ευρώπη σήμερα Είμαστε τρεις φορές πιο οικονομικά αποτελεσματικοί από το CNN και πέντε φορές καλύτεροι από το BBC. Αυτό κατέδειξε η ερευνά μιας, ε, του οικονομικού ελεγκτή ε, ότι είμαστε η πιο οικονομικά αποδοτική ιδιοσιογραφική επιχείρηση σήμερα για τα φαρσί. Ε, σας επιβεβαιώνω ότι πράγματι ο λόγος ε, χρήσης ε, της γλώσσα φάρση μόνο στο διαδίκτυο είναι δημοσιονομικός. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα την ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα πολύ καλά. Είπατε για ποιο λόγο επιλέξαμε τα Ουκρανικά, τα φάση και τα Αραβικά. Τα Ουκρανικά διότι ο Ουκρανό εταίρο σταμάτησε τη χρηματοδότηση. Έχουμε δηλαδή μια σύμβαση με τον εταίρο και ο εταίρο σταμάτησε τη χρηματοδότηση. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε την σύμβαση αυτή χωρί τον εταίρο. Ε, οφείλεται λοιπόν στη χρηματοδότηση από μέρου του εταίρου. Το ίδιο ισχύει για τα φάρση. Για τα περσικά, διότι είχαμε και εκεί έναν εταίρο, τι ε, εξωτερικέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποφάσισαν να μειώσουν τη χρηματοδότηση. Οπότε χρειάστηκε να βρούμε κάποιον άλλο ε, χρηματοδότη, κάποιον άλλο τρόπο μάλλον παραγωγή, διότι ήταν και έτσι αποδεχτήκε αδύνατο να διατηρήσουμε τηλεοπτική μετάδοση σε φάρση δεν ήταν δική μας επιλογή, δεν το αποφασίσαμε. Αν αύριο ε, με τα τουρκικά ο εταίρος ε, ε, για την τουρκική τηλεοπτική εκπομπή σταματήσει τη χρηματοδότηση, θα χρειαστεί να διακόψουμε και τα τουρκικά. στο λεπτό που μου απομένει, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ. Πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια παρανόηση, παρεξήγηση, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες κύριε Πρόεδρε και ζητώ να ζητήσω συγγνώμη Ίσως να είναι τα ανεπαρκή αγγλικά μου. Ήθελα να πω, εσείς μου δώσετε την ευκαιρία, αυτό είπα, μου δώσετε την ευκαιρία να εξηγηθώ, να σε εξηγήσω, να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεστε εδώ. Το σέβομαι. Ε... και το εκτιμώ ιδιαίτερα. αλλά δεν θέλω να λαμβάνω λάθος κατηγορίες, ψευδείς κατηγορίες. Δεν αναφερόμουν για αυτό εδώ το μέρος. Ε, δεν, δεν ακούστηκαν εδώ, δεν επαγγελθήκαν εδώ οι κατηγορίες. Ξέρετε, τους τρεις-τέσσερις τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλές κατηγορίες ε, κατά ημών και ε, θα τους ε, κυνηγήσουμε δικαστικά. Ε, δεν αναφερόμουν όμως εδώ σε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα να υπερασπιστώ την Euronews και να δώσω κάποιες εξηγήσει σε όλους εσά που φυσικά ε, παρακολουθείτε την Κρόνιος με τη δέουσα προσοχή όπως κάνετε τα περασμένα χρόνια. Οπότε ζητώ συγγνώμη για την παρεξήγηση αυτή. Δεν ήταν πρόθεσή μου. Um, uh, Ο κύριος Αμπαμόντε, πολύ σύντομα. Δεν απάντησα στο ερώτημα του κυρίου Μόργαν για το πόσα χρήματα κόστησε το Euronews τα τελευταία 10 χρόνια. Θα του ε, αποστείλω την απάντηση γραπτός. Το ερώτημα ήταν σημαντικό. Γιατί μας ρωτήσατε αν οι ελεγκτές ε, ρώτησαν, εξέτασαν το θέμα για την εξαρτησία μας. Στην αξιολόγηση που έγινε το 2014. Σημαντικό, έτσι. Η υποστήριξη του Euronews από το 2010 μέχρι το 2016 ήταν ε, από 19,5 εκατομμύρια ως 24,8 εκατομμύρια το 2016 με πικ το 2016, το 2012, συγγνώμη. Η αξιολόγηση των ελεγχτών ήταν ότι το Euronews κάνει περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι ο έλεγχος δεν ήταν οικονομικός έλεγχος. Κοίταξαν οι ελεγκτές όλα τα θέματα της συμφωνίας, της συμφωνιστερικής σχέσης την ευρωπαϊκή προοπτική, την πολυγλωσία, κοίταξαν, έθεσαν θέματα βιωσιμότητας του μοντέλου. Δεν αμφισβήτησαν καθόλου όμως ούτε την ανεξαρτησία ούτε την ευρωπαϊκή προοπτική. Επομένως, ναι, εξέτασαν όλα αυτά τα θέματα, εξέτασαν το κύριο θέμα της ανεξαρτησίας και δεν υπήρχε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Το να κάνει κανείς περισσότερα με λιγότερα δεν αποτελεί βεβαίως ε, ένδειξη ή δείκτη για την ποιότητα. Ε, έτσι ήθελα να το πω και αυτό. Ε, φτάσαμε στο τέλος της κοινής μας συνεδρίας. Να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε για κάποιες τελικές παρατηρήσεις και συνέχεια θα συνεχίσουμε εμείς με το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκρέσλε. Θέλω απλά να πω ότι το ε, ερώτημα θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε ε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση φώτισε ορισμένες διαστάσεις του ζητήματος, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Αν άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη, θα πρέπει να μας απαντήσουν ε, γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτε, τον κύριο Αμπαμότε και τον κύριο Γκαριμπέρτη για την παρουσία τους εδώ, για το γεγονός ότι απάντησαν στις ερωτήσει μας. Η Επιτροπή Πολιτισμού και αυτή από την πλευρά της θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρο της προσοχής της αυτό το θέμα. Σας ξαναευχαριστώ για την παρουσία σας.